Ladies and gentlemen, let's start. Thank you very much for coming. I must say, Mr. Butikova has less charisma than... Πρέπει να πω πως ε, ο κύριος Μπιουτικόφερ έχει λιγότερο χάρισμα από μένα. Α, ξέρω, ξέρω πως θα το, το ήξερα ότι θα το λέγατε. Λοιπόν, έχουμε κάτι το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο έκθεση Χέρμαν Φανρόμπο για τη Σύνοδο Κορυφής. Και επειδή βεβαίω ε, είναι ζητήματα προπολογισμού ενδιαφέρουν. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ μόνο με τους καλύτερους, με τους παρόντες. Και ε, νομίζω πως θα γίνει καλή συζήτηση. E Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας. Σας καλωσορίζω όλες, όλους και όλες. Έχουμε ειδικού εδώ πέρα. Ας ακούσουμε λοιπόν την καθηγήτρια Φιλομίνα Μαρή, ένα κλασικό αρχαιοελληνικό όνομα βλέπω διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Μέχρι πρόσφατα ήταν επισκέπτης καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο της ε, Μπρίζ και έχει είναι, τη μοναδική έδρα Ζαμονές στην Αυστραλία. Μετά έχουμε τον δόκτωρα Γιώ Λαϊβέη, διευθυντής του Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σιγκαπούρη. Ε, η οποία εκτός από καθηγήτρια στο της Ικαπούρης είναι και ερευνητής ε, διεθνών σχέσεων. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και μετά ο Δόκτωρ Γιώναθαν Χόλσλαγκ. Μόλις ήρθε με τα τρακτέρ εδώ πέρα. Και διδάσκει στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών ε, και είναι ερευνητή για κινέζικα ζητήματα. Νομίζω πως είναι σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί βεβαίως ασχολείται με το ζήτημα του μέλλοντος και για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο που θα έχει στην παγκόσμια τάξη λόγω παγκοσμίων τάσεων γιατί βεβαίως η σχέση αυτή έχει όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική σημασία. Άρα πρέπει να δούμε τι ρόλο θα παίξει η Κίνα και άκουσα πως τώρα προσγείωσαν για πρώτη φορά τζετ δικής τους κατασκευής σε αεροπλανοφόρο μια συμβολική ημερομηνία βεβαίως και από πλευράς ε, ασφαλείας ε, και οικονομικών. Γιατί βεβαίω ε, μια περιοχή και στον ελευθερό εμπορίο έχει και άλλα κίνητρα πέρα από το οικονομικό. Οπότε έχουμε πολλά ερωτήματα, πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω λόγο στην κυρία, στην καθηγήτρια Μαρή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ ε, εν μέσω ημών. Αυτή την ευκαιρία μου δίνεται για την ακρόαση και ιδίω για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο διότι το διδακτορικό μου αφορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση ήμουν βοηθό κάποιου βουλευτού στο παρελθόν. Οπότε γι' αυτό σα λέω είμαι ενθουσιασμένο που ξαναβρίσκομαι εδώ. Πριν από 20 χρόνια είχε πει κάποιο ότι η Ευρώπη έχει ελευθερία και τα πλούτη όμως τα έχει η Ασία. Λίγο αυτό ακραίο είναι, λίγο υπερβολή, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι συνομιλητές μα, επομένως ανέκαθεν είχαν διαφορετικά κανόνες, συνήθειες και όλα αυτά επομένως ε, βγαίνουν και στη σχέση μαζί τους και τώρα έχουμε ε, τις τεκτονικές αλλαγές ε, όσον αφορά την εξουσία, τη δημοκρατία, το εμπόριο και διαφορετικά είδη ασφαλείας. Οπότε τώρα συνεργαζόμαστε ε, ε, όσοι είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε αντίπαλοι, αλλά είμαστε και αλεξαρτώμενοι. Αλλά πάνε επί, επί επίσης και επίσης και στις πολυμερείς ε, συμφωνίες είμαστε μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συνέπεια, για να μπορέσουμε να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με τους Ασιάτες. Θα πρέπει να τους δείξουμε ότι έχουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι συνεπές, ότι έχει συνέχεια, το ίδιο ισχύει και για την ηγεσία της, αλλά και επίσης το ίδιο ισχύει και για την προσέγγιση της. Από την άλλη μεριά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αυτούς που έχουμε απέναντί μας στο τραπέζι. Ότι το σκηνικό στην Ασία δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Υπάρχουν πάρα πολλά δίκτυα συμμαχιών, δεν είναι γνωστό, δεν είναι εξαφέ Ποιοι είναι οι βασικοί συνομιλητέ εκάστοτε από την άλλη μεριά. Και οπότε το, το, το, το οποίο επομένως είναι πολύπλοκο, πολυμερές και το θέμα δεν είναι μόνο οι ελεύθερε συμφωνίε εμπορίου, ε, αυτές που τώρα περνάνε από διαπραγμάτευση, αλλά τα εργασιακά, τα, τα κλιματικά, οι δημόσιες συμβάσεις, η προστασιμότητα στις, στις κρατικές αγορές, ε, αλλά επίσης και το ότι, το ότι ολοένα και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πλησιάσει τα θεσμικά όργανα ε, της, της Ασίας όπως την συνάντηση κορυφής. Και γι' αυτό όμως θα πρέπει και εμείς να αποδείξουμε ότι ε, δεν έχουμε σχέσεις ε, υπερδυνάμεων αλλά εταίρων, συνομιλητών και αυτά θα πρέπει να είναι ιδέα Οπότε έχουμε κάτι το πολιτικά πολύπλοκο σαν σχέση αλλά έχουμε επίσης και κάποιες ιστορικές αντιφάσεις. Και εμείς ε, θα πρέπει κάτι να προσφέρουμε, που δεν μπορούμε να προσφέρουμε βέβαια την περιφερειακή ασφάλεια. Πάντως είμαστε πάρα πολύ δυναμικοί όσον αφορά την μη παραδοσιακή ασφάλεια, δηλαδή τις ε, πανδημίες, δηλαδή την ε, αρρωγή, όπως αφορά κάποιες ειρηνευτικές αποστολές και μετακινήσεις πληθυσμών, αλλά βοηθούμε και όσον αφορά την διατροφική ασφάλεια. Οπότε, ακόμα και αν εμείς θεωρούμεθα ως οικονομικός παίκτη, οι, πρωτοπόροι, οι πρωτοπόρες δράσεις είναι ανεπτυξιακή βοήθεια και παραδοσιακή και λιγότερο παραδοσιακή ασφάλεια. Οι άλλες προκλήσεις είναι ε, η εξή συμμετρία αλλά και και, η επαφή σε επίπεδο κορυφής. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμμετρία. Θα πρέπει να δούμε τους συνομιλητές μας ως ίσους και ότι έχουν και εκείνοι ε, τον ρόλο τους στην ισορροπία της περιοχής. Αυτό αφορά και τα, τα, τα συμφέροντα τα αμερικανικά επί στην περιοχή, αλλά και στα ε, διεθνή φόρα. Και έτσι μπορούμε να να αντισταθμίσουμε τις ΗΠΑ, να τις ανταγωνιστούμε εκεί. και ταυτόχρονα έχουμε τις, ε, ε, σχέσεις αυτές που είχαμε τη συνάντηση του Ιουλίου, ήταν πάρα πολύ ε, χρήσιμο αυτό και βέβαια θα πρέπει να δούμε το πώς δεν θα ταυτίζονται οι θέσεις μας με τις θέσεις των, των ΙΠΑ. Άρα θα πρέπει έτσι εμείς να κινηθούμε ε, σαν ένας ε, ενδιάμεσος σε συμφωνίες και δεν θα πρέπει επομένως να ταυτιζόμαστε με τις ΙΠΑ. Επίσης, συμμετρία αποτελεί και το ότι θέλουν οι συνομιλητές μας να υπάρχει περισσότερη εκπροσώπησή τους στα διεθνή φόρα ή ας πούμε να υπάρχει περισσότερη παρουσία τους, ανάμειξή τους στα της Γενικής Διευθύνσεως 20. Πάντως ε, υπάρχει συμμετρία και όσον αφορά το, το κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή το, ε, το κοινωνικό κράτος ε, είναι κάτι το οποίο διαφέρει για τους Ασιάτες. Το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, έχουν διαφορετικές απόψεις. Οι συνομιλητές μας επίσης. Συμμετρία υπάρχει όσον αφορά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος για τις περιφερειακές ρυθμίσεις και νομοθεσία. Και γιατί ε, εκεί ε, η ευρωπαϊκή, ε, η ευρωπαϊκή πλευρά αναπτύσσει επιχειρηματικότητα, αλλά δεν είναι πάντοτε το ίδιο ε, καλοδεχούμενη. Οπότε, όσον αφορά την ασφάλεια και την ε, ειρνευτική διαδικασία, ε, μπορούμε κάτι να κάνουμε, μπορούμε να έχουμε κάποιου είδου θεσμικέ δραστηριότητε, διότι έχουμε τη διαπεριφερειακότητα και επομένω έχουμε τέτοιε δυνατότητε, όπω έχουν και οι συνομιλητέ μα. Οπότε, για να μετρώ τώρα το άλλο θέμα, τη σχέση επίπεδο κορυφή. Θέλουμε να εκπροσωπούμε σε, σε, και εμεί σε, περισσότερα φόρα εκεί. Ε, πρέπει όμω να δεσμευτούμε και να αποδείξουμε ότι αξίζουμε ως συνομιλητή με του θα πρέπει επομένω να αποδίδουμε σημασία στον συνομιλητή, θα πρέπει να εμφανιζόμαστε, να είμαστε παρόντες αλλά το θέμα είναι ποιο εμφανίζεται, με, τι προσέγγιση, με τι ατζέντα που να έχει ε, συνοχή, λογική, συνέπεια. Ε, οπότε ε, επομένω χρειάζεται να έχουμε επαφή, χρειάζεται να έχουμε επαφή σε αυτό το ενότοτο επίπεδο εκεί που υπογράφονται αυτές οι συμφωνίες ελευθερού εμπορίου και άλλες ε, συμφωνίες ε, και σε επίπεδο ΑΣΕΑΝ στο βαθμό που θα ευδοκιμήσει. Και να δούμε τώρα κατά πόσον χρειάζεται μια καινούργια στρατηγική. Ε, είναι τόσο διαφορετική η Ασία που χρειάζεται να έχουμε πολλές στρατηγικές, όχι μόνο μία στρατηγική για την, για την Κίνα. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι πολιτικές που όμως δεν θα θεωρούνται ότι είναι κοινοτικές πολιτικές. Ε, είμαστε δωρητές, ας πούμε μετά το τσουνάμι ε, είχαμε βοηθήσει, αλλά αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται περισσότερο. Άρα θα πρέπει το μήνυμα να είναι πιο σαφές. Και θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στα συζητούμε τα δικαιώματα. Από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να τους βλέπουμε αφιψηλού, ε, να, να ότι είμαστε υπερόπτες ή ότι έχουμε αποκειοκρατικό ή μετα, απεικιοκρατικό ε, ύφο. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικές εμπειρίε που μπορεί να τι μεταλαμπαδεύσει, αλλά βέβαια ε, ενεδρεύει ο κίνδυνο του να θεωρήσουν ότι, είμαστε σνόμπ και ότι μόνο, κατ' εμάς, μόνο το ευρωπαϊκό μοντέλο ολοκλήρωσης ισχύει. Θα πρέπει να έχουμε να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα της Ευρωζώνης, αλλά θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούν να στηριχτούν σε εμά, ότι ε, μπορούμε να δεχτούμε ως εταίρους και όχι ως αντίπαλη δύναμη τους Ασιάτες στα, στα ε, τραπέζια των ε, διαπραγματεύσεων όπου θα πρέπει βεβαίως στον Ασιά να έχουμε έναν πρέσβη κάποιον δηλαδή που ασχολείται μόνο και αποκλειστικά με τα θέματα του Ασιαν και να μας αντιπροσωπεύει στην Τζακάρτα. Τώρα που έχουμε την ε, υπογραφή της συνθήκης για συνεργασία με την Άσιαν, τώρα έχουμε ε, τον λόγο να έχουμε κάποιο τέτοιου είδους εκπροσώπηση, να έχουμε κάποιο σύμφωνο διακυβέρνησης, δημοκρατικό, με ε, κάποιες αρχές που αξίζει να τις μοιραστούμε τους ε, άλλους μας τέλους εκεί, τους συνομιλητές, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Ιαπωνία, για παράδειγμα, να δούμε ε, τι, τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτά τα οποία είχαμε πει το 2001, ότι δηλαδή έχουμε και τη διάσταση αυτή της Ασίας που θα πρέπει να μην την ξεχνούμε ποτέ. Το δε πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ακούγεται με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται συνέπεια, πολιτική, στρατηγική, συνέχεια, συνοχή. Χρειάζεται να έχουμε επίσης ε, ενιαία προσωπικότητα και να ξέρει τέλο πάντων ο συνομιλητής ποιος θα εμφανιστεί για να συνομιλήσει, ε, τι ισχύει με την Προεδρία και κάθε φορά να είναι γνωστό ποιος και τι ρόλο έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να αναγνωριστεί ο διαφορετικός ρόλος των συμμάχων μας ε, να συνεργαστούμε στενά με κάποιες χώρες όπως η Αυστραλία και όπου τώρα ε, κατοικώ και σε αντίθεση με τις καθημερινές γραμμές του Ιουλίου που αφορούν τη ασφάλεια και θέματα εξωτερικής πολιτικής ο σχετικός ε, αιώνα, αυτό το, το, το, το έγγραφο για την Ασία, ε, αυτό που έχει ε, εκπονήσει η αυστραλική πλευρά, είναι ένα έγγραφο 300 σελίδων που μας δείχνει ότι θα πρέπει και εμείς να αντλήσουμε περισσότερο τις προκλήσεις που υπάρχουν και τα, τα ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα για την Ασία, να μάθουμε περισσότερο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια αλλά και σε επίπεδο επιχειρηματιών και επιχειρήσεων για να έχουμε επομένω περισσότερη συνεργασία όπως γίνεται και με τις σχέσεις μας με τις ε, ΕΠΑ. Μια άλλη πλευρά τώρα είναι το ότι υπάρχει μια ομάδα Ευρωπαίων που είναι ασιατικής καταγωγής αλλά έχουν ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είναι επομένω τέλεια αυτή η ευκαιρία. Μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτούς που απλά γλώσσας, κουλτούρας, ε, κοινωνίας ε, ξέρουν την Ασία. Αυτούς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ε, προς όφελός μας. Και έτσι να προχωρήσουμε σε αυτή την σχέση με τους Ασιάτες συνομιλητές. Επίσης, θα πρέπει μέσω αυτού του συμφώνου διακυβέρνηση είπα, να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποια φόρα συνάντηση στο ΑΣΙΑΝ και εδώ στην Ευρώπη. Εκεί θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι όπως ας πούμε την ε, ειρηνευτική διαμεσολάβηση, ε, τη βοήθεια για ε, διεθνωτικές μειονοτικές διαφορές, ε, που τα ξέρουμε αυτά από την Ευρώπη, ας πούμε να βοηθήσουμε στο ανάλογο εθνοτικό πρόγραμμα που υπάρχει στην Μπούρμα. Και έχουμε τις συμβασίες του εμπορίου, έχουμε εταιρικέ σχέσεις, διάφορες ε, συμφωνίες που έχουμε χρησιμοποιήσει, γιατί πάρα πολλά, το σκηνικό συνεχώς αλλάζει από το 1994 και μετά που έχουμε την νέα στρατηγική. Επίσης, ε, έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τον ρόλο των, των Αμερικανών, Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο, θα πρέπει να καταλάβουμε περισσότερο το ασιατικό ε, χώρο και ε, να δούμε το ότι χρειάζεται να υπάρχει συμμετρία, να μιλούμε σεμνά και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το, το καρότο και όχι το μπαστούνι όπως λένε στις επαφές μας να είμαστε συνεπείς στις εμπορικές ε, επαφές. Να αποδείξουμε ότι έχουμε αρχές και ηθική και να προσέξουμε διότι δεν, ε, δεν θα πρέπει να υπάρξουν ε, παρεξηγήσεις, να θεωρηθεί ότι είμαστε υπερόπτες. Απλώς να είμαστε μια ε, ευγενής βελούδινη δύναμη και έτσι να μπορέσουμε κι εμείς να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπαμε, τους Ευρωπαίους ασιατικής καταγωγής. Επίσης να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε τις μη κυβερνικές οργανώσεις που δρούν και εδώ στο Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά μπορεί να εμπλακεί και έχει ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τα ζητήματα διακυβέρνησης. Πολύ σημαντικό αυτό. Πρόκειται για μία ήπειρο που προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες. Όμως χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερο. Οπότε για να δούμε τι μήνυμα μπορούμε να στείλουμε στην Ασία. Μήνυμα συνέπειας, συνοχής, ε, παραδοχής των προβλημάτων της ε, Ευρωζώνης και πρόκειται για κάποια πρόκληση που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μαζί με τους Ασιάτες φίλους. Τέτοιο μήνα θα πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε τι, τι, τι άλλες προκλήσεις ε, έχει αυτού του είδους η σχέση με την άλλη επαφή του, την άλλη όχθη του ειρηνικού. και να δούμε πώς θα βρούμε κοινό έδαφος με τους συνομιλητές της άλλης Είναι πάρα πολύ πυκνό το σκηνικό εκεί από διαφορετικούς εμπλεκομένους. Και το θέμα δεν είναι μόνο τι θα γίνει, τι κάνουν στην Ανατολική Ασία, να δούμε τι κάνουν και οι Αμερικανοί, να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος της Ινδίας. Δεν υπάρχει επομένως μία και μόνη προσέγγιση η στρατηγική. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο μήνυμα δέσμευσης το οποίο να στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα ο δόκτωρας ή δόκτωρ Γιώ Λεϊχβή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καλέσατε για να μιλήσω. Το Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζουμε, με την συνθήκη της Λισαβόνας έχει ευρύτερο ρόλο να παίξει σε διάφορες πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής και πιστεύω ότι για μια πλήρη δέσμευση για την Ασία ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου είναι σημαντικός. Χρειάζεται, όπως είπε και η Φιλομένα ήδη, στην παρουσίασή της, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε κάθε επίπεδο. Όταν μιλάμε για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασίας, μοιάζει λίγο με το πουκάμισο, το πολύχρωμο που φορά, με πολλά ε, ζωηρά σημεία, αλλά εάν ε, κανείς ε, εργάζεται και δουλεύει εδώ σε αυτό το κλίμα των Βρυξελών, δεν αρκεί ένα πολύχρωμο πουκάμισο, χρειάζεσαι κάτι παραπάνω. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ασία έχουν αυξήσει τη συνεργασία μέσω διαφόρων ε, βάσεων ε, και ε, έχουμε ας πούμε τον ε, διαπεριφερειακό διάλογο ανάμεσα στην Ένωση και στην Ασία. Ε, έχουμε την Ευρωασιτική Συνεδρίαση, την ένατη η διάσκεψη έγινε στο Λάος πρόσφατα και βέβαια διάφοροι διμερείς διάλογοι γίνονται με βασικούς εταίρους Ασιάτες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία. Ωστόσο, τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα εξακολουθεί να υπάρχει μια αίσθηση πως η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΥΣ δεν έχει φτάσει στη στο πλήρε τη ε, δυναμικό και πρέπει να γίνουν περισσότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Νομίζω πως δεν έχουμε συμφιλειωθεί με τις διαφορές μας, με τις ασυμμετρίες που, για τις οποίες μίλησε η Φιλομένα και ότι ο διάλογος που έχει γίνει μέχρι στιγμής ε, βασικά εστιάζει την προσοχή στη ε, ρητορία και όχι στην ουσία. Αν θέλουμε να έχουμε μια δυνητικά καρποφόρα και θερμή και ε, σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία, πρέπει να έχουμε μια πιο μακρόπνοη άποψη και να υιοθετήσουμε μια θετική και ρεαλιστική στάση και προσέγγιση στο διάλογο και τη συνεργασία. Γιατί λέω, μιλάω για μακρόπνοη ε, ε, εικόνα ή άποψη. Χρειαζόμαστε τέτοια εικόνα γιατί παρά όλα τα λαϊκιστικά που λέγονται για το ότι παρακμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τη μεγάλη οικονομική δύναμη. παραμένει σταθερά στο 30% περίπου η, συνολική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα η Ασία αυξάνεται και αναπτύσσεται στην οικονομία αλλά και σε άλλες πτυχές. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να συνεργαστούμε. Και αυτό σημαίνει μια μακρόπνοη και βιώσιμη εταιρική σχέση με εμπιστοσύνη και ρεαλισμό. Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να γίνει ένας διάλογος μεταξύ ίσων. Αυτό το τόνισε η Φιλομένα, ότι δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε μία στάση υπεροπτική ανωτερότητας, ε. μια, μια, ένα διάλογο ίσως προς ίσως ε, για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε για τις διαφορές μας και να χειριστούμε τις αντιλήψεις μας. Αυτό που είναι σημαντικό στις σχέσεις αυτές είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις αντιλήψεις, ε, τις προτεραιότητες του καθενός, ε, όχι να προσπαθήσουμε να τις εξαφανίσουμε, αλλά να διαπραγματευτούμε για αυτές. Θα συνεχίσουμε να, έχουμε διαφορές. Το πώς θα τις ε, εξομαλύνουμε είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης και πρέπει επίσης να είμαστε ξεκάθαροι στις προσδοκίες μας. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι περιμένουμε δηλαδή από αυτή τη συνεργασία. Πιστεύω πως γίνονται τεράστιες αλλαγές στην Ασία και στην Ευρώπη καθώς και παγκοσμίω. Και οι δύο περιοχές αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις. Η Ευρώπη με το κρίση του χρέους, με τις δημογραφικές προκλήσεις. Στην Ασία έχουμε αυξανόμενη ανισότητα και πολλά άλλα προβλήματα. Ο κίνδυνος είναι επειδή πιστεύουμε πως έχουμε ο καθένας τα δικά μας προβλήματα να απομονωθούμε περισσότερο. Ε, και να παραμελήσουμε τον άλλον και να μην προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Γιατί πολλά από αυτά τα προβλήματα στην ουσία είναι αλληλένδετα. Πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις είναι και πλέον η ώρα να δούμε και να αναγνωρίσουμε την εξάρτησή μας και να επανεξετάσουμε το πώς θέλουμε να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε μια ισχυρή και σταθερή συνεργασία. Η Ασία και η Ένωση θα πρέπει να γνωρίζουν την πολυμορφία και την περιπλοκότητα, την ιστορία και τους θεσμούς που μπορεί να ορίσουν τις και τις προσδοκίες μας. Η Ασία μπορεί να μην έχει ακόμα μια συλλογική φωνή. Η περιοχή είναι ε, πολύ μεγάλη, ε, ε, διαφοροποιημένη και περίπλοκη και υπάρχουν διάφορες, διάφοροι οργανισμοί όμως νομίζω το ΑΣΕΑΝ είναι η πιο, πιο βασική δομή που υπάρχει και αποτελεί όλο ένα και πιο σοβαρό εταίρο στο μόνιμο παιχνίδι σχεδιασμού του μέλλοντος της Ασίας. Μπορεί να βλέπετε ότι κάποιες στιγμές επικρατεί ακόμα και αμηχανία αλλά, μέσα στο ΑΣΕΑΝ, αλλά παραμένει ο πιο σημαντικός οργανισμός, η πιο σημαντική δομή αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία μέσα σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ ίσων. Η Ένωση θα πρέπει να ακούσει και να προσπαθήσει να καταλάβει τις ε, τις ε, αντιλήψεις, τις προσδοκίες, ε, να διατυπώσει τις επιθυμίες και όχι να αναμειχθεί σε εκλογικούς νόμους, προδιαγραφές, αρχές κτλ. Να δηλώσει τα συμφέροντά της και τα ενδιαφέροντά της, να καταλάβει τις προτεραιότητες και να διαπραγματευτεί για τις διαφορές ώστε να βρεθεί κοινή, κοινό έδαφος και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τόσο η, το ΑΣΕΑΝ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζονται λιγότερο στα λόγια και να είναι πιο ανοιχτή στο διάλογο και να διαπραγματευτούν αυτέ τι διαφορέ, να χειριστούν τι διαφορετικέ προσδοκίε. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν και ακούγονται διάφορε φωνέ στην Ασία, μια βασική προσδοκία για την Ασία είναι να προσπαθήσει να λύσει τα κοινά, ε, να δει μάλλον ότι είναι κοινό συμφέρον να αναλυθούν τα προβλήματα του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προβεί σε βήματα κοινά μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να συνεργαστεί η Ασία, να σταθεροποιηθεί η παγκόσμια οικονομία και να αντιμετωπιστεί η πτυτικότητα των αγορών. We common in working together, Επίσης, ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε στην αναζήτηση πιο βιώσιμων ε, μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ε, άνευ απασχόλησης ανάπτυξης, της μεγάλης ανεργίας. Η αντιμετώπιση και ο διάλογος για τέτοια προβλήματα κοινωνικής οικονομίας πρέπει να γίνει μέσα από συνεργασία, να αναπτυχθούν καθολικές προσεγγίσεις, λύσεις, ακόμα και πριν από το σύστημα της εκπαίδευσης, της παιδείας, ώστε οι νέοι να μπορέσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που χρειάζονται στον, στην νέα πραγματικότητα. Πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία στον τομέα της ε, παιδείας, της των επιστημών, ε, γιατί υπάρχει αλληλεξάρτηση και διαβρώνεται η δυνατότητα των κρατών, ακόμα και των περιφερειών, ολόκληρων περιφερειών να λειτουργήσουν απομονωμένα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Μπορεί να σκεφτόμαστε ότι μονάχοι μας αντιμετωπίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι ε, αλληλένδετες. Με αυτό το, το μήνυμα κλείνω την επισήγησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον Τζόναθαν Χόλσλεκ. Ευχαριστώ κύριε Μπιουτικόφερ. Στη σύντομη παρουσίασή μου, εγώ θα ήθελα να προτείνω τρία επιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφεληθεί πάρα πολύ από την άνοδο της Ασίας. Δεύτερον, δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο πως θα βελτιωθεί η κατάσταση στα επόμενα χρόνια. Και ο καλύτερος τρόπος και αυτό είναι το τρίτο μου επιχείρημα, είναι να έχουμε μια εντονότερη πολιτική ε, γειτονίας ε, και μια πιο μικρή πολιτική Ασίας. Ε, μπορεί να μην ακούγεται σωστό κοτσόψιος, αλλά νομίζω πως ισχύει. Ας δούμε πρώτα απ' όλα τι κερδίσαμε από την Ασία την τελευταία δεκαετία. Κάθε χρόνο πάνω από 100 εμπορικές αποστολές Πηγαίνουμε στην Ασία, έχουμε γύρω στα 650 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν επενδυθεί στην Ασία, αλλά αν δούμε συνολικά το εμπορικό ισοζύγιο, που εξακολουθεί νομίζω να αποτελεί σημείο αναφοράς, φαίνεται πως ακόμα έχουμε μείνει σε μια ελληματική σχέση παρά το κάποιο επενδυτικό εισόδημα και την αύξηση του εμπορίου. Βλέπουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ελληματική εμπορική σχέση με την Ασία. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Κίνα. Ε, πέρα από τρεις χώρες έχουμε ελληματικές σχέσεις με όλες τις ασιατικές αγορές και οικονομίες. Όταν μιλάμε για διεθνή συνεργασία, νομίζω πως δεν έχουμε μία σύγκληση από πλευράς ε, κανόνων πέραν από την Ιαπωνία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ φαίνεται πως διαφέρουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για προτεραιότητες και ε, φιλοδοξίες στην παγκόσμια πολιτική όσον αφορά την στρατηγική εταιρική σχέση με μεγάλες παίκτες όπως η Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία. Δεν υπάρχει πολλή ουσία από πλευράς ε, συνεργασίας ασφαλείας ε, και μεγάλων διεθνών προκλήσεων. Ένα τρίτο ζήτημα, αν δούμε μια δεκαετία σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Ε, αν συγκρίνουμε γενικά τις απόψεις ε, χωρών της Ασίας την περίοδο 2010-2012 με την περίοδο 2006-2008 βλέπουμε πως οι απόψεις ε, της Ασίας έχουν επιδεινωθεί όσον αφορά την Ευρώπη. Δεν έχουμε τώρα το χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά θεωρώ πως ο απολογισμός μιας δεκαετίας ε, ε, εταιρική σχέσης Ασία-Ευρωπαϊκής δεν είναι πολύ ενθαρρυντικός. Τι μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν από το μέλλον. Εγώ θεωρώ πως η Ασία πηγαίνει σε ένα μέλλον με αναταράξεις και θα πρέπει να περιμένουμε, ε, όπως είπα, αυτές τις αναταράξεις. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα τα όρια της ανισόρροπης ανάπτυξης. Εάν δούμε παραδείγματος χάρη την οικονομική κατάσταση της Κίνας, υπάρχει λόγος ανησυχίας οπωσδήποτε, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει καμία συνένεση για το πώς θα, δούμε, θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισορροπίες. Δεδομένου δε το ότι η υπόλοιπη Ασία εξαρτάται από αυτή την αναξιόπιστη, το αναξιόπιστο κινητήρα ανάπτυξη. Βλέπουμε πω οι πολιτικέ ελίτ σε διάφορε ασιατικέ χώρε έχουν μπροστά του ε, κοινωνικέ αναταραχέ και ζητήματα νομιμοποίηση. Το άλλο ζήτημα βεβαίω είναι η ισορροπία ισχύω. Το ανέφεραν και οι ομιλήτριε. Η άνοδο τη Κίνα ε, απαντάτε με μια τάση ισορρόπησης ε, και τη τείχος αντίδραση της Κίνας. Γιατί θεωρώ πως αυτό είναι λόγος ανησυχίας. Γιατί δεν θεωρώ δεδομένο πως η ψύχρεμη προσέγγιση που υφίσταται ακόμα στη στρατηγική σκέψη και τη διπλωματία της Ασίας παρά τα κάποια ε, ναυτικά επεισόδια ε, μπορεί να μην συνεχιστεί αν υπάρχει οικονομική και κοινωνική ε, αστάθεια και μπορεί να υπάρχει και μια στρατηγική αν θέλετε αμφισημία δηλαδή συνεργασία αλλά και αυξανόμενο εθνικισμό. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Για μένα δέκα βασικές προκλήσεις υπάρχουν. Δεν μπορώ να επεκταθώ τώρα. Αλλά νομίζω πως η πρώτη αξίζει κάποια περισσότερη προσοχή. Πρώτα απ' όλα οι ανερχόμενες δυνάμεις, η Κίνα και η Ινδία, έχουν την τάση να ε, ασκούν έναν οικονομικό εθνικισμό και δεν έχουν καμία τάση να πάνε προς την κατεύθυνση του ανοίγματο ε, και των ε, θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων. Αυτό χωρίς μια πολιτική, οικονομική αυτοπεποίθησης μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Και αυτό το οποίο επίσης θεωρώ πως ε, αξίζει λίγα λόγια παραπάνω είναι η πολυμέρεια. Η αποτελεσματική πολυμέρεια είναι βασικό κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής μας, αλλά βεβαίως επειδή υπάρχει ακόμα μία δυσαρμονία με τους ε, ασιάτες εταίρους μας, δεν ξέρω κατά πόσον ταυτιζόμαστε σε όλα τα ζητήματα. Τα υπόλοιπα δεν θα τα αναφέρω, ίσως αν μου κάνετε ερωτήσεις να επεκταθώ. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν για τη χάραξη τη πολιτική τη Ένωση. Νομίζω πω σημαντικό είναι να έχουμε τι σωστέ προτεραιότητε. Οπωσδήποτε η Ασία δεν είναι η μόνη περιοχή η οποία ζητάει την ε, προσοχή μα, αλλά οπωσδήποτε θεωρώ πω ε, πρέπει να υπάρξει κάποια χάραξη στρατηγικής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίζουμε τις αξίες μας με συγκεκριμένες σκληρές, αν θέλετε, δυνατότητες. Προαπαιτούμενο νομίζω για να είμαστε αξιόπιστος εταίρος είναι η οικονομική ανάκαμψη, νομίζω πως αυτό έχει ουσιαστική σημασία, στρατηγική σκέψη όπως είπα και οι δύο πρώτες ομιλήτριες ε, έκαναν πολύ σημαντικές συστάσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για την πολιτική, πρώτα απ' όλα είναι ένας ε, συνδυασμός ε, αύξησης του ωφέλους και μείωσης των κινδύνων. Τι σημαίνει αυτό, όπως είπα, μια πολιτική εμπορική πιο στιβαρή. Επίσης πρέπει να εξυπηρετήσουμε τις νέες πόλεις της Ασίας. Υπάρχουν πολλές νέες σημαντικές αγορές. Και πολύ εξαγωγήση λοιπόν στον τομέα των υπηρεσιών. Επίσης για τις συνεργασίες, ειδικά στα χαρτιά ε, είναι σαφείς αυτές οι απτήσεις, αλλά όταν μιλάμε για τη διατήρηση των διαλόγων πρέπει να υπάρχει ένα παιχνίδι δύο επιπέδων καθώς ειδικά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει δυνατότητα συντονισμού με τα κράτη-μέλη και μπορεί νομίζω να καταστήσει σαφές το τι μπορεί να προσφέρει και μετά περνάμε στις ανάγκες ασφαλείας της Ασίας. Προφανώς πολλές ασιατικές χώρες μας ζητάνε να εμπλακούμε στις ε, θαλάσσιες διαφορές τους ε, για να στηρίξουμε παραδείγματο χάρη ε, κάποιες ρυθμίσεις. Σημαντικό είναι λοιπόν πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε και την περιφέρειά μας. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε σε διάφορες περιφέρειες αυτό το οποίο μας ρωτάνε οι διπλωμάτες και επισημαίνει τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για εμάς για να την ε, θαλάσσια ασφάλεια στον κόλπο του Άντεν, ε, ε, στην τρομοκρατία, στη Δυτική Αφρική, όπου πολλές ασιατικέ χώρες έχουν επενδύσεις. Τι γίνεται με τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Δεν βλέπουμε την Ευρώπη πουθενά. Νομίζω λοιπόν πως και οι ασιατικές ανάγκες στον τομέα της ασφαλείας βρίσκονται στη γειτονιά μας και αυτό νομίζω πως πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα. Μετά, ένα εναλλακτικό σχέδιο να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ε, δική μας ε, την ε, ευαλωτότητα. Δηλαδή κάποιες χώρες ε, οι οποίες ε, εξακολουθούν να έχουν μόνιμα πλεονάσματα. Ένα άλλο ζήτημα είναι πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις προδιαγραφές ε, προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να προωθούμε υψηλότερε πράσινες προδιαγραφές και κοινωνικές προδιαγραφές παρά το ότι συχνά έχουμε αντίσταση από τις ασιατικές ε, πρωτεύουσες. Και το άλλο ζήτημα που είναι μακροπρόθεσμο αφορά τις εισαγωγές ε, πρωτογενών ε, αγαθών, καθώς αναμένεται πως οι εξαγωγές της Κίνας μεταλλευμάτων θα αυξηθούν την επόμενη δεκαετία, έχει κρίσιμη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία να καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να μειώσουμε την έκθεσή μας στις ε, αγορές εμπορευμάτων, οι οποίες είναι, έχουν πολλές ανακατατάξεις. Και τέλος, πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε και εμείς μοχλούς πίεσης και βεβαίω έχουμε και το ζήτημα της οικονομικής ανάκαμψης. Αυτό είναι το φλέγον ερώτημα που ρωτάνε όλοι στην Ασία η Ευρώπη. Θα, θα ξεπεράσει την κρίση. Νομίζω πως πρέπει να δούμε πως ε, είμαστε σε κάποια παρατεταμένη παρακμή, οπωσδήποτε αυτό θεωρούν πολλοί Ασιάτες. Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και αξιολόγησή τους τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης, ε, της αντιστάθμισης της Κίνας για να έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια και τέλος όπως είπα θεωρώ πως θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροή. αν μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην σταθερότητα της γειτονιάς μας. Δηλαδή αυτή η ζώνη ανασφάλειας από την Βαλτική, τη Μέση Ανατολή μέχρι το Γιβραλτάρ. Σημαντικό λοιπόν για να τα δούμε όλα αυτά από μια παγκόσμια προοπτική για μένα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τη γειτονιά μα. Θα μπορέσουμε λοιπόν να ασκήσουμε πίεση στις σχετικέ δυνάμει μόνο εάν καταφέρουμε να γίνουμε απόλυτα απαραίτητη δύναμη στι γειτονικέ μα χώρε. Ευχαριστώ. So very much, Jonathan. Σας ευχαριστώ και εγώ. Jonathan και έτσι φτάνουμε στο τέλος των ε, τριών ε, εισηγήσεων και στο τμήμα ερωταπαντήσεων αυτή τη ακρόασης και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ το προνόμιο της Προεδρίας και να ε, θέσω κάποιες ερωτήσεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα τρομερά από όλες τις παρουσιάσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Απλά να επανέλθω σε κάποιες από αυτές. Να ξεκινήσω με ένα σύντομο ανέκδοτο από την τελευταία διάλογο στην Σαγκριλά όπου βασική ομιλία έγινε από τον πρόεδρο της Ινδονησίας και σε εκείνη την ώρα των ερωταπαντήσεων του ρώτησε ο συντονιστής από την CSIS κατά πόσο πίστευε πως η Ευρώπη και η Ρωσία θα έπρεπε να παίξουν ένα ρόλο στην θέματα ασφαλείας της Ανατολικής Ασίας. Και η απάντηση του Ινδονήσιου Προέδρου ήταν βεβαίω η Ρωσία πρέπει να παίξει ρόλο. Τελεία. Εσείς ε, μιλήσατε για προσδοκίες. Πέρα από την επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων της Ευρώπης, τι προσδοκίες μπορεί να υπάρχουν για την Ευρώπη η πρόταση που μόλις παρουσίασε ο Τζόναθαν Χόλσλακ ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο φροντίζοντας κάποια από, τα ευρύτερες, από τις ευρύτερες ασιατικές βλέψεις παγκοσμίω θα μπορούσε να είναι αυτός ένας ρόλος. Και μια δεύτερη ερώτηση προς εσάς. Υπάρχουν καλά παραδείγματα κρατών μελών που να παίζουν ένα πιο δραστήριο ρόλο από ό,τι άλλα και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή δράση ώστε δηλαδή ως Ένωση να βασιστούμε στο τι έχουν ήδη κάνει ή κάνουν κάποια Και προς τον δόκτωρα Μάρε μιλήσατε για την Ευρώπη ως μια πιθανή δύναμη εξορρόπησης. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μάρς πάντα θα περιμένει, ο Άρης συγγνώμη, περιμένει την ε, Αφροδίτη για να είναι ισορροπημένος. Αλλά, με πάση περιπτώσει, σε έναν τέτοιο ρόλο η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει κάποια φιλοδοξία. Γιατί η δήλωση στην οποία εσείς ε, αναφερθήκατε για την κοινή δήλωση ανάμεσα στην ε, Χίλαρη Κλίντον και τη Λέδη Άστον προσπάθησα να το βρω κάπου στα μέσα της Ευρώπης και δεν το βρήκα ούτε σε μία εφημερίδα ούτε σε μία τηλεοπτική εκπομπή. Πώς θα παίξει έτσι εξισορροπητικό, ρόλο η Ευρώπη. Ίσως μπορούσατε λοιπόν εδώ να επεκταθείτε και επίσης θα με ενδιέφερε να δώσετε κάποιες ε, αποσαφηνήσεις όσον αφορά αυτό το σύμφωνο διακυβέρνησης και τη διάσταση της επιχειρηματικής κοινότητας στο πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στην Ένωση και στην Ασία. Και για σένα, Τζόναθαν, η αλλαγή της άποψης των Ασιατών για την Ευρώπη. Η εκτίμηση για την Ευρώπη ήταν καλύτερη από ό,τι ε, πριν από δύο χρόνια, μόνο στην Νότια Κορέα όμως. Αυτό στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ή συμβαίνει κάτι άλλο. Και έπειτα, και οι τρεις σας αναφέρατε τον αγώνα εξοπλισμού που γίνεται στην Ανατολική Ασία και το ρόλο που παίζουν ορισμένες ε, χώρες, ε, κράτη-μέλη της Ένωσης, σε σχέση με τις εξαγωγές τους προς την περιοχή. Ίσως μπορείτε λοιπόν να το αναλύσετε περισσότερο. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο για όποιον θέλει να θέσει ερωτήσεις. Ας απαντήσετε πρώτα όμως αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ όσον αφορά για την ερώτησή σας. Τι προσδοκίες υπάρχουν ε, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς τι, τι θεωρούμε σαν έναν ε, πάρα πολύ σημαντικό ε, οικονομικό παράγοντα. Και αυτό είναι η μέρη μας. Θέλουμε να ε, συμβάλλει στην επίλυση, να αντιμετωπίσει την κρίση τέλο πάντων η Ευρωπαϊκή να μπορεί να συμβάλλει περισσότερο. Σα βλέπουμε σαν οικονομικό παίκτη, αλλά επίση διαπιστώνουμε ότι επίση και σε μη ε, παραδοσιακές πλευρές της ασφάλειας και εκεί είναι σημαντικός ο ρόλος σας. Ε, το είπε η Φιλομίνα και επίσης. Ε, είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο περιφερειακό φόρουμ του ΑΣΕΑΝ είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την πολιτική διπλωμάτη Συμβάλλει σημαντικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την, την, την ανάπτυξη δυνατοτήτων για αντιμετώπιση προβλημάτων με προληπτική δημοκρατία για διατήρηση της ειρήνης, για επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων ε, σε διάφορες ε, ε, αποστολές του ΟΑΣΕ. σε διάφορα φόρα επομένω σε όλα αυτά τα σημεία υπάρχουν επαφέ και οπότε έχουμε και εμεί αυτό το επίπεδο προσδοκίε και επίση δεν θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας ανταγωνιστή, τον είπα. Γιατί είστε σε, άλλη διάσταση και οικονομική ισχύς, νομοθετική, ε, κανονιστικής φύσης, εκεί δηλαδή που ξέρετε τα θέματα και εμείς έχουμε να μάθουμε από σας. Θα πρέπει και εμείς να μάθουμε, να υιοθετούμε κάποια πρότυπα, να, να δανειστούμε από εσά την εμπειρία για αυτά τα οποία γνωρίζετε. Να, μερικά από τα ζητήματα τα οποία είχα να σας αναφέρω. Και εδώ βάζω τελεία. Σας ευχαριστώ, κυρία Μάρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι ο εξισορροπητικός ρόλος είναι το ατού, το φόρτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και η σας Δεν έχετε εσείς τον 7ο στον ειρηνικό. Αυτό όμως είναι πλεονέκτημα από πολλές πλευρές. Σίγουρα πολλοί εκεί πέρα αντιπαθούν τη είπα αλλά μπορεί να μην σα ξέρουν, αλλά δεν, δεν σα αντιπαθούν εσά εκεί πέρα. Οπότε δεν, δεν είναι το θέμα τη ε, παραδοσιακή ε, ομπρέλα ασφάλεια. Ε, δεν είναι αυτό ο ρόλο σα και άρα αυτό που είναι ο ρόλο σα να το εκμεταλλευτείτε με θετικό τρόπο. Γιατί τι έγινε με του Αμερικανού, ιδίω επί Μπού, θεωρούν το αντιμουσουλμάνοι οι, ε, οι Αμερικανοί ε, χάλασαν οι σχέσεις ε, με την Ασία λόγω της, της πολιτικής του Λευκού Οίκου. Εσείς δεν περάσετε από τέτοια δεσσαραστή φάση, υπάρχει ο διαπολιτικός διάλογος και επομένως έτσι να είστε ήρεμοι, δύναμοι, αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό. Οπότε, έρχομαι και στο δεύτερο θέμα. Το θέμα του συμφώνου διακυβέρνηση. Τι θα πει καλή διακυβέρνηση, παρά την κρίση που σοβεί στην Ευρώπη. Υπάρχει σωστή διακυβέρνηση, γίνονται σεβαστά ανθρώπινα δικαιώματα και ε, ακόμη ε, υπάρχει αντιπάθεια προς την διαφθορά. Ε, οι κυβερνήσεις υιοθετούν σε πολιτικές κατά της διαφθοράς και αυτό δεν είναι χρήσιμο για την Ασία, για τις δημοκρατικές χώρες. Ε, και σε αυτό, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να υπάρξει ε, και μέσω του διαλόγου Σαγκριλά τέτοιου είδους ε, επαφή για το κράτος δικαίου κλπ. Το κράτος προνοίας, να, το, το, πάντοτε προσφέρουμε στους ταξιτζίδες να μάθουμε που, τι, τι θέματα υπάρχουν και είπαν ότι ακριβώς υπάρχει δυσφορία γιατί δεν υπάρχουν ρυθμίσεις και κράτος προνοίας ε, γιατί στην Ευρώπη την άλλη μεριά υπάρχει μεγάλη ποικιλία μορφών καπιταλισμού, υπάρχει σεβασμό για του ε, μη προνομιούχου. Να τι θα πει καλή διακυβέρνηση. Και τέλο, όσον αφορά τη ρυθμιστική νομοθεσία, ε, η Ασία όντω προσβλέπει, γιατί εδώ, εδώ επίση είναι ένα φόρτε των Ευρωπαίων. Αυτό αφορά και το διάλογο της Ασίας με τον ΠΟΕ, οπότε και σε αυτό το σημείο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι υπεύθυνη, κοινωνική, ε, πολιτική διακυβέρνηση. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να αρχίσει ο διάλογος με τις δημοκρατικές ασιατικές δυνάμεις. Επίσης, ε, όσον αφορά τους επιχειρηματικούς κύκλους, και εκεί υπάρχουν πολλές δυνατότητες ε, στην πλατφόρμα του ΑΣΕΑΝ ΑΣΕΑΝ συν η Νότια Κορία, Κίνα, εκεί είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιο είδους όργανο να υπάρξει κάποιο δίκτυο να υποστηρίζονται έτσι οι ευρωπαϊκές εταιρείε που θέλουν να ε, ασκούν εμπορία ε, στην Ασία. Αυτές οι αντιπροσωπείες ε, που έχουν και εμπορικό ακόλουθο θα μπορούν να έχουμε διάλογο της επιχείρησης προς επιχείρηση και εκεί να εξηγείται γιατί είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει προσβασιμότητα στις ε, κρατικές ε, προμήθειες και διαγωνισμούς, τι γίνεται με, τα, με, με την ε, πνευματική ιδιοκτησία. Τώρα, όσον αφορά τους εξοπλισμούς, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενισχυτικό. Θα πρέπει και αυτό εδώ να το κοιτάξουμε τι γίνεται. οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το εμπάργκο των όπλων. Άρα είπαμε να εκμεταλλευτείτε τα πλειοκτήματα της ε, η Ευρώπη, να ε, κοιτάξει τι θα γίνει με τους πρόσφυγες, γιατί υπάρχει σημαντική ε, εμπειρία για μετακινήσεις πληθυσμών κέντρο Τζακάρτας, για την συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου, Πολλέ πολλές δυνατότητες υπάρχουν σε, αυτά τα επίπεδα που νομίζω ότι ακόμα δεν τι έχουμε εκμεταλλευτεί. Ξεκινήσαμε όσον αφορά το τι γίνεται στην Κορέα και ήταν πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι υπήρχε μια εξελικτική διαπραγματευτική διαδικασία και όσο προχωρούσαμε στα συμπεράσματα είδαμε ότι εκεί ε, τα πράγματα δεν πήγαιναν γραμμικά όσον αφορά το τι μπορούσαμε να πετύχουμε. Τώρα, το άλλο ερώτημα που αφορούσε του εξοπλισμού, την κούρση των εξοπλισμών, αυτό πολύ σοβαρό. Το θέμα δεν είναι μόνο ο εξυγχρονισμό των ενοπλών δυνάμεων, είναι η αύξηση. Η αύξηση, ε, ε, το, το, μεγάλο των, στόλων η, η Κίνα τώρα να φυγεί πολύ περισσότερα πολεμικά πλοία από ό,τι είπα και γενικά όλο ένα και περισσότερο εξυγχρονίζεται ο στρατός σε όλη την ευρύτερη περιφέρεια. Και συμφωνώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το πού πουλάμε όπλα. Προσοχή, επομένω. Ε, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσει το εμπάρκο στα όπλα. Όσο γίνεται να προσέχουμε. Και γιατί εκτός από την ε, Κίνα να προσέχουμε και την Ινδία. Γιατί πολλές φορές είναι το ίδιο ε, φιλοπόλεμη ας πούμε ή ε, όσο και η Κίνα εις βάρος της ε, Σρι Λάγκα, εις βάρος του Μπαγκλαντές. Τέλος πάντων, είχε γίνει μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα ε, κάποιων υπευθύνων του ναυτικού και λέγανε ότι σε κάποια ώρα της Ασίας πρόκειται να ε, κατασκευαστεί ένα ναυπηγείο. Και ξέρω ότι αυτό δεν, δεν αφορά μόνο μία εταιρεία. Ναυπηγείο για να εξυπηρετεί γύρω-γύρω. Επομένως, μπορείτε τώρα να δείτε το ότι χρειάζεται να υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Δεν είναι σημειακό το θέμα μόνο όσον αφορά το εμπάργο της βάσης της Για την εφικτή ισορροπία τι προσδοκούν από εμάς οι Ασιάδες. Δεν είναι τόσο σαφές. Πολλές φορές έχοντας στις Βρυξέλλες να... και επιζητούν κάποια δήλωση για την ε, θάλασσα της Κίνας, αλλά χρειάζεται κάποιο είδους συμβολική υποστήριξη για τις διαπραγματεύσεις. Θέλουν την Ευρώπη για να αποκτήσουν ακόμα ε, ακόμα μια αγορά, ε, να μην την αφήσουν μόνο στους Κινέζους. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι θέμα ισορροπίας αυτό, είναι θέμα του να χαλαρώσει η πίεση. Δεν μπορούμε να αυτό ε, να το εξισώσουμε, ούτε καν να το συγκρίνουμε το ρόλο των Αμερικανών. Και μην υπερεκτιμούμε τη μόχλευση που μπορούμε να, να, να ασκήσουμε, να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά την διάσταση των όπλων, θυμάμαι μια νέα φράση που διάβασα, που μάλλον θα είχε πει ο Walter Russell Mead, που μίλησε για στρατιωτικό κενσιανισμό. Αλλά... Αλλά θέλω να δώσω και την ευκαιρία στους παριστάμενους να κάνουν ερωτήσεις, ε, παρατηρήσεις ναι. Ε, κτλ. Αν οι βουλευτός λοιπόν θέλουν να πούν κάτι οπωσδήποτε, αλλά και οποιοδήποτε άλλος αν θέλει να λάβει το λόγο, παρακαλώ συστηθείτε, κάντε τις ερωτήσεις σας και πείτε μας σε ποιον ε, απευθύνεστε. Ποιος θέλει λοιπόν να μιλήσει πρώτος. Παρακαλώ. Δεν βγαίνετε από το τμήμα πολιτικής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω μια ερώτηση για το ζήτημα αυτό της ρόψης. Ε, ε, μιλάμε για εξισορρόπηση της επιρροής των ΙΠΑ αλλά τον Ιούλιο η Βαρόνη Άστον και η Υπουργό η κυρία Κλίντον εξέδωσαν μια κοινή δήλωση για την συνεργασία Ασίας Ειρηνικού. Οπότε δεν ε, εξισορροπούμε πλέον γιατί έχουμε διαλέξει μια πλευρά και ακολουθούμε την προσέγγιση των ΙΠΑ, οπότε δεν τίθεται ζήτημα εξισορρόπησης να μάθω λοιπόν ποια είναι η αντίληψη εντό του ΑΣΙΑΝ για την κοινή αυτή δήλωση, Πώ το είδαν οι διάφορε κυβερνήσει. Ευχαριστώ. Άννα Γκόμες. Με συγχωρείτε μόλις ήρθα γιατί είχαμε, είχαμε την διάσκεψη των Προέδρων για το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Ναι, ναι, μου το εξήγησε ο Έλμαρ και έχασα τις παρουσιάσεις οπότε ίσως κάνω μια ερώτηση που έχει ήδη απαντηθεί. Αλλά θα ήθελα να γνωρίζω τις απόψεις σας ε, για τις συνέπειες ε, της αύξησης ε, στρατιωτικής δύναμης της Κίνας για ολόκληρη την Ασία και την Ευρώπη. Δεν μιλάω μόνο για τις οικονομικές συνέπειες αλλά και την αύξηση σε σχέση με τις ε, πιθανές συγκρούσεις. Πώς το βλέπετε αυτό να επηρεάζει τις λοιπές σχετικές φορές. Έχουμε άλλη ερώτηση. Then we uh, start uh, with a round of answers. Please. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις απαντήσεις. Παρακαλώ λοιπόν. Ναι. Θεωρώ όταν οι κυρίες Κλίντον και Άστον έκαναν την κοινή δήλωση για την Ασία ειρηνικό, θέλω να ομολογήσω πως δεν πρόσεξαν και πολύ. Αλλά ταυτόχρονα, κατά την άποψή μου, γιατί εγώ το, το είδα, σκέφτηκα δεν είναι καλό σημάδι αυτό, γιατί σκέφτηκα θα ακολουθήσουν η ίπα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει την και εμείς ακριβώς όταν είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούμαστε περισσότερο με την οικονομική πτυχή ενώ από πλευρά ασφαλείας δεν έχει δική της ανεξάρτητη πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλουμε να το πάμε παραπέρα μπορούμε να πούμε πως ε, χωρίς να θεωρώ όλους ε, τους Ασιάτες ε, απλά ως ακαδημαϊκός ποια θα ήταν η αντίδραση, ότι δηλαδή η Δύση ενώνεται εναντίον της Ασίας. Ε, Αυτό σκέφτηκα όταν είδα τη δήλωση. Αλλά όπως είπα, θεωρώ πως στην πραγματικότητα, αν δούμε την κατάσταση στο επίπεδο της πολιτικής, δεν θεωρώ πως ε, υπήρχαν πολλές ε, αντιδράσεις στη δήλωση αυτή. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Ανεξαρτήτως του αν και κατά πόσον απασχόλησε τον τύπο αυτή η δήλωση, οπωσδήποτε θα εξετάστηκε. Με ενδιαφέρον στο, Βερολί... στο... στο Πεκίνο. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να διατηρήσει δηλαδή μια πιο ανεξάρτητη στάση, αναγνωρίζοντας την σημασία των είπα στην περιοχή. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά σε συγκεκριμένους τομείς, σε συγκεκριμένες πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένες λέω. Αυτό θεωρώ όμως πως ε, δεν την ενισχύει, αντιθέτω την υπονομεύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια ξεκάθαρη φωνή. Χρειαζόμαστε κάποιο λογισμικό αναγνώρισης φωνής. Οι συνέπειες επίσης της, ε, του ανταγωνισμού εξοπλισμών. Και το ζήτημα της ε, νότιας ε, θάλασσας Κίνας δεν θα εξαφανιστεί. Υπάρχουν και συνοριακές διαφορές και προκλήσεις. που οι λοιπές χώρες Ασίας θα το θεωρήσουν ως ένα μήνυμα πως πρέπει και οι ίδιες να εξοπλιστούν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προσεκτική και σε ποιον εξάγει, αλλά βέβαια να κοιτάει και τη σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ινδονησίας. Πρέπει να κοιτάει το τι συμβαίνει στις χώρες του Αζίαν και στην Καμπότζη, Βιετνάμ και Ινδονησία. Πρέπει να τα δούμε λοιπόν πολύ σοβαρά όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ναι, για την δήλωση Άστον Κλίντον. Αυτό το οποίο δεν μου άρεσε είναι το πώς προέκυψε. Προέκυψε από κάποια σοβαρή διαδικασία. Λάβαμε κάποιες προσκλήσεις από την Ουάσιγκτον και λόγω κάποιων έτσι προσωπικών φιλιών πήγαμε και κάναμε αυτή τη δήλωση. Το πώς το είδε η Κίνα ε, ήταν κάτι το αρνητικό και νομίζω πως ε, εξασθένησε θα έλεγα την εμπιστοσύνη που είχαμε στο Πεκίνο. Αυτό το οποίο ακούμε από τις άλλες χώρες περιοχής είναι πως και πάλι ήταν μία απόδειξη του γεγονότος πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ανεξάρτητη και πάλι ακολουθούσε τις είπα για το ερώτημα της κυρίας Κόμες για τους εξοπλισμούς της Κίνας. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Και εάν πάλι μιλήσετε με ανθρώπους στο Πεκίνο, που ξέρουν δεν βλέπουν καμία διάθεση υποχώρησης, αντιθέτως έχει αναγνωρίσει η κινέζικη ηγεσία πως ε, η Κίνα πρέπει να αποκτήσει ναυτικό ανοιχτή θαλάσσης, να έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τα συμφέροντά της στο εξωτερικό, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο να κατηγορούμε μόνο την Κίνα. Πρέπει να δούμε πως ε, πρόκειται για ένα δίλημα ασφαλείας με τις ΗΠΑ, κυρίως ε, καθώς υπάρχουν διαφορετικά στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Οι Αμερικανοί εδώ και δεκαετίες προσπαθούν να διατηρήσουν την ε, στρατιωτική τους υπεροχή στον δυτικό ειρηνικό και να έχουν μια περίμετρο ασφαλείας όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Ευρασιατική Ήπειρο. Και με βάση την ιστορική τους ε, εμπειρία οι Κινέζοι θέλουν να το αλλάξουν αυτό και θεωρούν πως ε, θα γίνουν όριμοι δύναμοι μόνο αν έχουν τουλάχιστον το επίπεδο ε, στρατιωτικών δυνατοτήτων όπως είπα στην περιοχή αυτή. Οπότε δεν ξέρω αν είναι κάποια επιθετική στάση από την κινέζικη σκοπιά είναι αμυντική. Αλλά το δίλημα αυτό νομίζω πως θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα όλων των συγκρούσεων στην περιοχή. Νότια, Ανατολική, θάλασσα της Κίνας. Για εμένα λοιπόν είναι κατά βάση το ζήτημα της ε, δυσπιστίας ε, που υπάρχει μεταξύ ε, Κίνας και ΙΠΑ. Πρώτα πρέπει να αποκτήσουν αυτοί οι δύο γίγαντες και οι γεμόνες μεγαλύτεροι εμπιστοσύνη μεταξύ του και μετά υπάρχει περιθώριο διαπραγματεύσεων σε ένα πολυμερέ ε, πλαίσιο. Και πάλι μετά νομίζω πως είναι κάτι το ε, δύσκολο το να βρει την ισορροπία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε πως ε, έχουμε και γεωπολιτικά συμφέροντα και φιλοδοξίες που δεν συμπίπτουν πάντα με αυτά τον είπα. Ευχαριστώ. Θα Σαμπίνε με πολιτική σύμβουλος των Πρασίνων. Εμείς ως ε, αντιπροσωπεία ΑΖΙΑΝ πριν από χρόνια βρεθήκαμε στα κεντρικά του ΑΖΙΑΝ και μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα και τότε ήταν σαφές πως αντιπαρέστε ε, αντίληψη την δική τους για το στρατιωτική και την ασφάλεια με την ευρωπαϊκή και την αμερικανική έλεγχη. Οι δικές μας χειρονίες δεν χρειάζεται να επενδύσουμε πολύ στο στρατό, το βλέπουμε αλλιώς. Ε, τώρα όμως όταν συζητάμε για τους εξοπλισμούς φαίνεται πως ακολουθούν την κατεύθυνση όλων των υπολείπων και δεν υπάρχει πλέον διαφορά. Κατόπιν είναι λυπηρό κατά την άποψή μου. Βλέπετε μια κάποια διαφορετική προσέγγιση. Είπατε πως δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να μιμηθούμε τις είπα εδώ πέρα, οπότε θα ήταν καλό να ακούσουμε πως ε, στον Αζιάν ε, ε, μπορεί ακόμα να σκέφτονται ενός διαφορετικού τύπου ασφάλεια. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο είναι πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Περισσότερο ε, για το Ιράν παρά ε, για την Παλαιστίνη. Νομίζω πως η παρατήρησή σας ήταν ενδιαφέρουσα παρά το ότι δεν συμφωνώ με την ανάλυση σας. Οι Ευρωπαίοι όσον αφορά τη στάση του προ το Ιράν. Και αν πάει κανεί στην Ινδονησία, το πρόβλημα μεταξύ Σουνιτών και Σιητών ε, μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες συγκρόσει Τη θέση της Ευρώπης στο Ιράν ή έχω λάθο. Και τέλο κλιματική αλλαγή. τελείω διαφορετικό θέμα. Δεν υπάρχει ένα τρόπο να ευθυγραμμιστούμε επ' αυτού. Ευχαριστώ. Είναι ο τελευταίος γύρος ερωτήσεων. Αν σκέφτεστε λοιπόν να, βάλτε, να θέσετε ερώτηση, το είναι η ώρα τώρα. Άννα Γκόμες, πάλι. Όσον αφορά την αντίληψη περί κρίσης στην Ευρώπη, Οικονομικής και Πολιτικής. Ποια είναι η εικόνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ε, τι είναι. Ένα εμπορικό κέντρο. Ότι όλα είναι στη φτύνια. Επίσης, εν ώψη του γεγονότος ότι η Ασία και πολλές ασιατικές χώρες επηρεάζονται από τις δικές τους ε, κρίσεις ε, που το το 70 αποκόμισαν ε, διδάγματα από εκείνη την κρίση και από την ε, παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Αντιμετωπίζουν τα θέματα που όλοι λέμε ότι αντιμετωπίζουμε, όπως π.χ. έλεγχο των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Η Σιγκαπούρη εξακολουθεί να θεωρείται από τις άλλες χώρες ως το πλυντήριο για την ε, σφοροδιαφυγή και τις απάτες, φορολογικές απάτες. Άλλος κανείς, παρακαλώ. Τερίζα Κόμπα από τη Γραμματεία της Επιτροπής. Μια μεγάλη διαφορά Ανάμεσα στη Δύση, τουλάχιστον την Ευρώπη και τις ασιατικές χώρες της διεθνής σχέσης, είναι η στάση απέναντι στην κυριαρχία σε σχέση με την ευθύνη την, ε, για προστασία, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και η πρόσφατη κρίση δείχνει πως αυτός είναι ένας βασικός λόγος μπλοκαρίσματος. Προχωρούμε προς ένα κόσμο πολλαπλών δυνάμεων. Η Ασία φαίνεται να εξελίσσεται ως προς αυτά, αλλάζει σε σχέση με αυτή την αντίφαση ανάμεσα στις δύο υπήρους. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Επανέρχομαι στο εμπόριο. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά ήθελε να διαπραγματευτεί μια περιφερειακή FTA με την περιοχή του ΑΣΕΑΝ. Για κάποιους λόγους που δεν έγινε αυτό και άλλαξε η πορεία. Και τώρα διαπραγματευόμαστε διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχει κάποια σκέψη στο ΣΕΑΝ ότι ίσως θα μπορούσε να ξαναλλάξει πορεία ή να αποδεχτεί αυτή η στρατηγική. Τζόναθαν, θες να αρχίσεις εσύ αυτή τη φορά. Η πρώτη ερώτηση όσον αφορά τις εξελίξεις για το ΑΣΕΑΝ και το κατά πόσο αυτό διαφέρει από τις άλλες περιφέρειες. Αν δεν νομίζω πως υπάρχουν διαφορές. Αν δούμε λοιπόν ποιες πλατφόρμες ε, ενισχύονται και σε ποιες πλατφόρμες δαπανούν τα χρήματά τους οι χώρες του ΑΣΕΑΝ, θα δούμε ότι δεν διαφέρουν από άλλες χώρες. Πολλές εντάσεις και τριβές ανάμεσα στην Κίνα και τις άλλες χώρες και τις χώρες του ΑΣΕΑΝ θα δούμε πως είναι πιο, σε πιο περιορισμένη κλίμακα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει τάση για βελτίωση και άμβληση αυτών των συγκρούσεων. Δεύτερη ερώτηση για το ρόλο της Μέσης Ανατολής σε σχέση με το Ιράν. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο θέμα και δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να εκτιμήσει, να αξιολογήσει δεκαετίες, τη δεκαετία της πολιτικής πώς αυτό γίνεται αντιληπτό στις Ισλαμικές χώρες για την Νοτιοανατολική Ασία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στην Ασία εν γέννη ισχύει το εξή ότι δηλαδή βασικά εμείς είμαστε ουραγοί της πολιτικής των ΗΠΑ προκειμένου να επιδιώξουμε τους δικό μας συμφέροντα και στόχους απέναντι σε χώρες όπως το Ιράν ίσως. Τώρα, χρηματοπιστωτική κρίση. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, ιδιαίτερα βέβαια όταν δούμε το Πεκίνο και πάμε και μιλήσουμε με τον κόσμο που δουλεύει εκεί μας ρωτάνε αν θα μείνουμε κολλημένοι στην κρίση για δεκαετίες. Να δούμε, πρέπει ωστόσο να δούμε αν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ή όχι την κρίση, να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι δεν θα χάσουμε πολλά χρήματα αγοράζοντας ε, ομόλογα πούμε από την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Όταν κανείς προχωρήσει περισσότερο στην συζήτηση, στην ουσία στρέφονται στον εαυτό τους. Λένε ότι εντάξει έχετε τα προβλήματά σας στην Ευρώπη και ότι παρά την πολιτική βαβούρα και τις σκέψεις κορυφής θα το ξεπεράσετε. Αλλά να δούμε εμείς, εμάς, εμείς τώρα πρέπει να εξορροπήσουμε την οικονομία μας και εκ νέου είμαστε αυτορχικό κράτος και μπορούμε να έχουμε πιο πολύ μόχλευση για την επιδίωξη οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά δέχονται πως το ίδιο πρέπει να γίνει και στις ε, ασιατικές χώρες και ότι είναι δύσκολη διαδικασία και για την Κίνα και για τις υπόλοιπες χώρες της Ασίας. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της αλεξάρτητης. Θεωρούν ότι είμαστε ευάλωτοι, αλλά αναγνωρίζουν πως και εκείνοι είναι πολύ ευάλωτοι. Και ότι βέβαια το επόμενο βήμα είναι να αξιολογήσουμε πόσο και σε ποιο βαθμό μπορεί κάτι τέτοιο να οδηγήσει σε μακροοικονομική συντονισμό, αμοιβαία στήριξη για την G20 και ευθυγράμμιση σε εκείνο το επίπεδο. Γι' αυτό το επόμενο βήμα δεν το βλέπω να γίνεται. Ξέρουμε πως είμαστε στην ίδια βάρκα. Αλλά από αυτό μέχρι που να φτάσουμε σε συντονισμό και στήριξη για παγκόσμια διακυβέρνηση έχουμε ακόμα απόσταση. Και τέλος, εδώ από τον συνάδελφο όσον αφορά την κυριαρχία και τις διεθνείς οργανισμούς. Οι περισσότερες ασιατικές χώρες όσον αφορά τις πολιτικές τους αξίες είναι, βρίσκονται εκεί που εμείς βρισκόμασταν στις αρχές του 20ου αιώνα. Δηλαδή δίνεται έμφαση στο ρόλο του κράτους, στα σύνορα, στον έλεγχο της κοινωνίας και νομίζω πως αυτό είναι φυσιολογικό και θα πάρει χρόνο να ξεπεράσει αυτές τις ιδέες η Ασία και να προχωρήσει κάπως στην αντίληψή της για αυτά τα πράγματα. Για τους διεθνείς οργανισμούς σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει προσεκτικά να παρακολουθήσουμε ναι, θα είμαι σύντομο. Ε, και όχι μόνο βλέπουμε πως υπάρχει μια τάση για συντονισμό ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ασιατικές χώρες και τα, τους διεθνείς οργανισμούς εις βάρος των δικών μας συμπερώντων, αλλά βλέπουμε και προσπάθεια των μεγάλων ασιατικών δυνάμεων να φτιάξουν δικά τους πολυμερή κανάλια, διάβλους με αφρικανικές, λατινοαμερικάνικες χώρες και έτσι πολύ συχνά ε, πιέζουν για αξίες ε, που είναι αντίθετες με τις δικές μας. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε όταν θα μιλήσουμε για διεθνή σχέση. Ευχαριστώ και τώρα για τον Δόκτωρ Γιάου. Ευχαριστώ να απαντήσω για την αυστριακή προσέγγιση για την ασφάλεια. Οι περισσότερες ε, ασιατικές χώρε θα έλεγα πως έχουν ένα συνολικό πλαίσιο ασφαλείας. Όχι όσον αφορά την ανθρώπινη ασφαλεία, γιατί το βλέπουμε από πλευράς ε, Κρατική ασφάλεια. αλλά είναι κάτι περισσότερο οπωσδήποτε από την άμυνα. Ε, γι' αυτό ακριβώς τονίζουμε ιδιαίτερα την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό ε, εξετάζουμε συνολικά το ζήτημα. και, Δουλεύω και πάω. Και ίσως πράγματι ο φόβος της Κίνας έχει οδηγήσει σε κάποιο σε κάποια αύξηση των εξοπλισμών. Τώρα, το πώς βλέπουν την τωρινή κρίση στην Ευρώπη. Αυτή είναι μας. Το βλέπουμε περισσότερο σε εξή ότι η κρίση στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την οικονομική κρίση. Είναι η κρίση του κοινωνικού συμβολέου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που είναι δύσκολο να επιληθεί. Γνωρίζουμε πως θα χρειαστεί καιρός και η οικονομική κρίση νομίζω μπορεί να επιληθεί. Αλλά ε, το ζήτημα του κοινωνικού συμβολέου είναι κάτι άλλο. Και ε, εδώ πέρα το αντιμετωπίζουμε αυτό και πολλές ασιατικές κοινωνίες ε, αυξάνεται η ανισότητα και κοιτάμε τις τροπίες μας και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όπως ε, είπα. Γι' αυτό ακριβώς τονίζουμε το ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλον, να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις πολιτικές και να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα, στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Βεβαίω, οι κοινωνίες διαφέρουν, έχουν διαφορετική ιστορία, κοινωνία, αλλά μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα και να ε, προχωρήσουμε προς ε, το μέλλον. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Εδώ από τον λόγο. κύριε σας ευχαριστώ. Δεν θα απαντήσω όλες τις ερωτήσεις, γιατί περισσότερες από αυτές έχουν ήδη απαντηθεί. Κράσεις, κρίσεις. Η κρίση ανέκαθεν βοηθούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει προς περισσότερη ολοκλήρωση. Άσιαν Συντρία, η πρωτοβουλία Τσαγμάη, μετά υπήρξε πολυμέρεια και βεβαίως η ανταπόκριση διέφερε, αλλά τα μαθήματα τώρα που αντλούνται είναι πολύ μας στην Ευρώπη και στο παρελθόν λέγαμε τι μπορεί να διδάξει η Ευρώπη, αλλά τώρα βλέπουμε τι μπορεί να διδαχθεί από την Ασία όσον αφορά την μετριοφροσύνη, όσον αφορά την συγκράτηση των δαπανών, όσον αφορά ε, τις ρυθμίσεις του τραπεζικού δικαίου. Τώρα όσον αφορά το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. υπεγράφη η συνήθεια εργασία με τον Ασιαν, αυτό σημαίνει και επίση και μη ανάμειξη. Όμως δεν ξέρω εάν χρειαστεί θα θελήσει να προστατεύσει τα κεκτημένα Ευρωπαϊκή Ένωση. και όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση, ε, ίσως προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ασία και Νότιο Ειρηνικό εις βάρος της, της ε, ε, εθνικής κυριαρχίας. Ξέρω ότι δεν το πάτε εκεί, αλλά θα παραμείνει σημαντική εθνική κυριαρχία ακριβώς λόγω των εδαφικών προστριβών που υπάρχουν Άρα βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν αντιφάσεις και πολυπλοκότητε. Για τις συμφωνίες ελευθερών εμπορία προχωράνε και εκεί η ατζέντα της Ένωση είναι πλούσια. Επίση, όσον αφορά τη συνδίκη με την Κορέα, αυτό σημαίνει ότι οι Ασιάτες συνομιλητές διαπίστωσαν ότι απέσπασε αξιόλογα πράγματα η Κορέα. Άρα αυτό είναι πλεονέκτημα για εκείνου που θα έρθουν να κάτσουν στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους για την ε, συμφωνία με τον Ασιαν. Αλλά βέβαια θα έχουν προηγηθεί με επιμέρους χώρες. Συμφωνίες όπως ας πούμε με την ε, Μπούρμα. Οπότε είναι, αυτό είναι περιφερειακή πολιτική επιλεκτική. Κάτι τέτοιο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ασκεί παράλληλα με τι ε, γενικότερε συμφωνίε και έχει τι διμερεί με επιμέρου χώρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα λέει το πρόγραμμα ότι, λέει ο Πρόεδρο, θα πρέπει να έχουμε τα, τα, την εξαγωγή συμπερασμάτων τώρα. Δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Απλώ να ε, συμπεράνω εγώ ότι ελπίζουμε να έχει συνέχεια αυτό ο προβληματισμό και ευχαριστώ του ε, τρει καλεσμένου μα γιατί πραγματικά μα ε, είπαν τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους και μας μάθατε πολλά. Παρακαλώ και εσείς να τους ευχαριστήσετε με ένα θερμό χειροκρότημα.